Σεπτεμβρίου λοιπόν θα ξεκινήσουν οι κυρώσεις αυτέ. Οι αρμόδιε Ιταλικέ αρχέ με ενημέρωσαν για την εκλογή του κυρίου Άντζελο Τσόκα από τι 7 Ιουλίου. Ο κύριο Τσόκα θα αντικαταστήσει τον κυρία Τζον Λούκα Μπονάνο και καλώ ορίζω λοιπόν τον νέο συνάδελφο και να σα υπενθυμίσω ότι πλέον συγκαταλάγεται και μάλλον ε, υποβάλλεται και πρέπει να υπακούει στον κανονισμό του Κοινοβουλίου και συμμετέχει ανάλογα στα όργανα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η νομική υπηρεσία, η νομική